επιχειρήσεων από τρίτα κράτη. Δεν θα δεχτεί δηλαδή τίποτε το οποίο να υπονομεύει το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έληξε η συζήτηση εδώ. Κύριε Επίτροπε. Σημείο στην ημερήσια διάταξη, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είναι δήλωση της Επιτροπής με θέμα χρήση κοινοτικών εμπορικών σημάτων στην εσωτερική αγορά. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Μπαρνιέ. Monsieur le Commissaire, vous avez la parole. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα εμπορικά σήματα έχουν ε, ουσιαστική σημασία στο σύγχρονο εμπόριο. Επιτρέπουν την αναγνώριση, την προέλευση των προϊόντων, των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας σταθερό επίπεδο ε, ποιότητας, προωθώντας την εικόνα των επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στο ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα είναι χρήσιμο για τις επιχειρήσεις μας και ένα μέσο να καταπολεμηθεί η Έχουν ληφθεί αποφάσεις οι οποίες θέλουν να περιορίσουν τη χρήση του, ευρωπαϊκού σήματος επικαλούμενες στις ε, απαιτήσει σύμφωνα τις οποίες η χρήση ενός εμπορικού ευρωπαϊκού σήματος σε ένα μόνο κράτος μέλος δεν θα αποτελεί ε, ευρεία χρήση αυτού του σήματος. Ευχαριστώ τους βουλευτές οι οποίοι επέσαν την προσοχή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή την κατάσταση την οποία παρακολουθούμε από πολύ κοντά διότι το πλεονέκτημα του Ευρωπαϊκού Σήματος είναι προσφέρει σε όλες τις επιχειρήσεις ακόμα και τις μικρομεσαίες ένα χρήσιμο εργαλείο για να προστατεύσουν το σήμα τους σε ευρωπαϊκό κλίμακα. Ο κανόνας βάσει του οποίου κάθε σοβαρή χρήση ενό κοινοτικού σήματος από τον κάτοχο αρκεί, ανεξάρτητα από τον χώρο χρήση της εντό της κοινότητας, θεωρήθηκε από όλου του χρήστε σαν ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του σήματος. Αυτός ο κανόνας είναι συνεπής με το ενιαίο χαρακτήρα του κοινοτικού σήματο και με τις αρχές της ενιαία αγοράς. Οποιοδήποτε νέος περιορισμός στη χρήση του κοινοτικού σήματο θα, θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την καταπολέμηση της παραποίηση, η οποία στο σχέδιο ΣΥΓΜΑΤΑΚ προβάλλει τη δέσμευση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της πειρατείας και της παραποίησης. Τι πρέπει να γίνει μπορούμε το κοινοτικό σήμερα, αποτελεσματικό μέσο όπως είπα για την καταπολέμηση παραποίησης διότι ε, παρέχει πλήρη ε, ασφάλεια προστασία σε όλη την επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα εξωτερικά της σύνορα. Τα παραποιημένα προϊόντα τα οποία εισέγονται μαζικά από τρίτες χώρες αυτή τη στιγμή πρέπει να μπορούν να κατάσχονται με βάση το, τις τε, τελων, κοινοτικές τελωνιακές διατάξεις στα σύνορα της Ένωσής μας κάτι τέτοιο θα μπορούσε να κάνει την πρόσβαση στο, στο κοινοτικό σήμα πιο δύσκολη για τις νέες επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν αρχικά σε, στο, στο εσωτερικό της χώρας τους και αρχίζουν τις εξαγωγές τους μόνο όταν αποκτήσουν κάποιο μέγεθος. Η δράση λοιπόν αυτών των επιχειρήσεων θα μπορούσε να καταστεί πιο δύσκολη αν δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν το κοινοτικό σήμα προτού διευρύνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Και υπάρχουν αυτό συμφωνεί με το πνεύμα πολλών πολιτικών των χωρών μας οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην πρόοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό επιβεβαιώνω κυρίες και κύριοι βουλευτές ότι οι υπηρεσίες μου θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη από πολύ κοντά. Έχουμε, αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν θα επικυρώσουν αυτές τις αποφάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την χρήση του ελληνικού σήματος ε, που παραβιάζουν τι αρχέ της ενιαίας αγοράς. Τώρα θα πάρουν το λόγο ομιλητές εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, η κυρία Χάντζλικ για ε, δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που μόλον ότι η ώρα είναι προχωρημένη είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό εμπορικό σήμα στην ιστορική αγορά. Είμαστε εμείς το ΕΛΚ που παρουσιάζει αυτή την πρωτοβουλία. που γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Επίτροπε, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους συναδέλφους στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και την ΙΜΚΟ. Το ΕΛΚ ήταν ανέκαθεν πεπισμένο πως η ιστορική αγορά συστάθηκε προκειμένου να καταργηθούν τα σύνορα ανάμεσα στα κράτη-μέλη και θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο για την κατάργηση των εμποδίων. Γι' αυτό λοιπόν προωθήσαμε την χρήση κοινοτικών εμπορικών σημάτων στην ιστορική αγορά. Χάρη σε αυτό το σύστημα εγγυόμεθα στις επιχειρήσεις μια ενιαία προστασία στον επικράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, ε, στην προστατευμένε ε, στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν ε, μας ανησυχούν κάποιες αποφάσεις που έλαβαν ορισμένοι οργανισμοί για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία ή των πνευματικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ακούσαμε κύριε Επίτροπε που πέτε ότι αυτές οι αποφάσεις βρίσκονται σε σύγκρουση με τι αρχές της εσωτερική αγοράς και την υπονομεύουν. Γι' αυτό η ομάδα μας ε, θα υποστηρίξει μια προσέγγιση η οποία θα προβλέπει και μιλάμε για την κοινωνική προσέγγιση που θα ε, αποτελεί εχέγγυ για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και σας ρωτώ, τι θα γίνει κύριε Επίτροπε αν η νομολογία των ε, κρατών μελών δεν συμφωνήσει με την θέση της Κομισιόν μήπως ε, δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού αναφορικά με τα εμπορικά σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσέγγιση των νομοθεσιών των ε, κρατών μέλων. Ευχαριστώ. Πολύ. Τώρα ο κύριος Ταραμπέλα εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών για δύο λεπτά επίσης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Σήμα εδώ και 16 χρόνια επιτρέπει την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης και υπαρκή προστασία για τον καταναλωτή, για την ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για υπηρεσία είτε για, που προσφέρει το προϊόν, είτε πρόκειται για το σήμα του. Το ίδιο αποβαίνει φίλο των επιχειρήσεων, μικρών και μεσαίων, όλων των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μα επιτρέπει να προχωρήσουμε, γιατί μέσα σε μια ιστορική αγορά μόνο ένα πραγματικό κοινοτικό σήμα επιτρέπει την αποτελεσματική προστασία. Το κόστο του είναι αρκετά χαμηλό και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για τι αρχέ επιτήρηση τη αγορά και των τελωνίων. Στις 14 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με μια αποφασή του λέει ότι χρειάζεται αποτέλεσμα τεχνικό για να μπορεί να καταχωρηθεί ως σήμα κοινοτικό ένα προϊόν. Αυτό σε απάντηση του αιτήματο της επιχείρησης Lego με τα τουβλάκια που ήθελε τα τουβλάκια της να το ε, προστατέψει με σήμα κοινοτικό. Και την πρόταση στο δικαστήριο. Και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε, ένα νέο κανονισμό, ε, έχουμε ανάγκη για ένα νέο κανονισμό, ο οποίο θα παρακολουθεί τι τεχνολογικέ εξελίξει, την παγκοσμιοποίηση εφενό και το ίντερνετ εφετέρου. Μην ξεχνάμε ότι στόχος μας πάντοτε είναι να προσφέρουμε πλήρε πληροφορίε, κατανοητέ και την επαρκή προστασία για τον καταναλωτή μέσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Των φιλελευθέρων, η κυρία Βίκστρομ έχει το λόγο για δύο λεπτά ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που σήμερα μπορούμε να έχουμε αυτήν την τόσο σημαντική συζήτηση, μόνο ότι η ώρα είναι ιδιαίτερα προχωρημένη. είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πως μας δίνει μεγάλες δυνατότητες για την κατάργηση των συνόρων και να ανοίξουμε τις, τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες και να μπορέσουμε έτσι να ευημερίσουμε ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Αυτό το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Η Ευρώπη δεν ε, μπορεί να προχωρήσει και να ενισχυθεί μόνο βασιζόμενη σε πολιτικές πρωτοβουλίες ε, και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πραγματική οικονομική ανάπτυξη βασίζεται στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα. Η Ευρώπη λοιπόν θα ανακάμψει, θα αναπτυχθεί εάν ε, ευημερούν οι επιχειρήσεις της. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία που να τις προστατεύει. Θα πρέπει σε εκ τούτου να καταργήσουμε τους φραγμούς στο εμπόδιο που παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ε, αφορά ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και πολλές φορές ε, η γραφειοκρατία τους κόβει τα πόδια. Εγώ λοιπόν ανέλαβα το έργο να επικρίνω τα κράτη-μέλη που ενεργούν ε, κατά των ε, κοινωνικών συμφερόντων και, κατά των ε, κοινωνικών εμπορικών σημάτων. Είναι απαραίτητο λοιπόν όλα τα αγαθά να προστατεύονται από εμπορικό σήμα στην εσωτερική αγορά. Το κοινωτικό εμπορικό σήμα κύριε Επίτροπε χρειάζεται να τύχει προστασίας. Ελπίζω σε αυτού του πως ε, η Ευρωπαϊκή Τροπή θα παρεύει για την προστασία του σε όλη την κοινωνική επικράτεια. Τρία λεπτά, κύριο Χάρμπουρ, από την ομάδα των ε, συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας μου και ως Πρόεδρος ε, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο πραγματικά γιατί κατέστησε απόλυτα σαφές ότι η συμπεριφορά των δύο ε, γραφείων στον Μπένελουξ και την ε, Ουγγαρία είναι παντελώς απαράδεκτες. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, διότι πρόκειται για επίθεση στι θεμελιώδει αρχέ τη εσωτερική αγορά. Και είμαι ικανοποιημένο για το γεγονό ότι όλοι οι ομιλητέ υποστήριξαν τι αποφάσει που θα λάβει ο Επίτροπο και η Επιτροπή για πρακτικούς λόγους. Είναι σύμπτωση εντυπωσιακή ότι αυτά τα δύο γραφεία ε, εμπορικών σημάτων εδρεύουν ε, στη χώρα της τωρινής και της επόμενης προεδρίας εγώ θα φροντίσω όταν ο Υπουργό Εσωτερική Αγορά έρθει στην Επιτροπή μου και ο Ούγγρο Υπουργό από τον Ιούριο, Ιανουάριο και πέρα, θα του υποβάλουμε αυτό το ερώτημα και θα του ζητήσουμε να απευθυνθούν στα γραφεία εμπορικών σημάτων και να πούν ότι αυτό είναι απαράδεκτο, διότι αποτελεί ουσιαστική επίθεση στις βασικές αρχές της, της εσωτερικής αγοράς που απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση κατά εταιριών, κατά επιχειρήσεων οπουδήποτε λειτουργούν σε μια ενιαία αγορά. Και σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα διότι αυτή η πρόταση, η προτινόμενη δράση εάν εφαρμοστεί θα δημιουργεί διακρίσεις εναντίον των μικρών επιχειρήσεων διότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που θα επηρεαστούν κυρίως από μια τέτοια απόφαση, διότι μπορεί να καταχωρήσουν ένα νέο εμπορικό σήμα για ένα προϊόν σε όλη την επικράτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας μια επανάσταση, εντυπωσιακή επανάσταση στην εσωτερική αγορά με, με, και έναν θαυμάσιο τρόπο προστασία των σημάτων. Μπορεί να χρειαστούν πέντε χρόνια για να κυκλοφορήσει το προϊόν του στην αγορά. Και τι θα ανακαλύψουν όταν θα πάνε στην Ουγγρική αγορά, ότι το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων τη Ουγγαρία καταχώρησε αυτό το εμπορικό σήμα σε μια άλλη επιχείρηση. Κάτι το απαράδεκτο. Μετά από τόσο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μα για την εναρμόνιση τη ενιαία αγορά, να έχουμε αυτά τα δύο γραφεία εμπορικών σημάτων καταχώρηση εμπορικών σημάτων να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Το κόστος καταχώρησης ενός ε, κοινοτικού σήματος έχει μειωθεί σημαντικά και αυτά τα δύο γραφεία προσπαθούν να διατηρήσουν το καθεστώς και να επιτρέπουν σε άτομα να καταχωρούν εμπορικά σήματα στην δική τους επικράτεια. Πρόκειται για ίδια συμφέροντα τα οποία πρέπει να καταπολεμήσουμε διότι αντιβαίνουν στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπονομεύουν, όπως πολύ σωστά είπε ο Επίτροπος, μια ουσιαστική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι η καινοτομία, η κυκλοφορία νέων προϊόντων στην αγορά και να καταστεί πιο αποτελεσματική ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάρμπουρ. Έχουν ζητήσει δυο συνάδελφοι να παρέμβουν στη συζήτηση. Η κυρία Ροϊτόβα, καταρχάς. Για ένα λεπτό παρακαλώ, κυρία Ροϊτόβα. Eh, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Και με χαρά ακούω ότι μέσα στον χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει την ε, νομοθεσία για το Ευρωπαϊκό Σύμμα με απλούστευση και πιο, πιο χαμηλό κόστος. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ακόμη ένα μέσο για την αντιμετώπιση των παραποιημένων προϊόντων. Επίση, με χαρά ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται να ενσωματώσει και τη δική μου πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής προστασίας για το ευρωπαϊκό σήμα. Γιατί δυστυχώ ε, το σήμα ποιότητας, ποιότητας και ασφάλειας, το οποίο θέλουμε να προστευθεί, ε, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πολλών ε, καταχρήσεων η προστασία του σήματος, CE δηλαδή, θα πρέπει να, να είναι ισοδύναμη με ποιοτικά προϊόντα για τον καταναλωτή και να προστατεύει τον ε, παραγωγό από την, ε, τον αθέμητο ανταγωνισμό. Η προστασία αυτή δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος γιατί είναι απλώς δυνατόν η καταχώρηση των υπηρεσιών, της υπηρεσίας του Αλικάντε μπορεί να επεκταθεί και για να καλύψει αυτό το θέμα. Βλέπω ότι ομόφωνα όλοι συμφωνούμε πως ε, η επέκταση του κοινοτικού σήματος αποτελεί φυσική συνέπεια της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας προϊόντων και σημάτων. Δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν κανείς να διαφωνεί με τους στόχους αυτούς. Γι' αυτό θα πρέπει κάθε δυνατή κύρωση να επιβληθεί προς τα κράτη εκείνα που ε, απειθαρχούν και να ε, μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να τα πείσουμε να συμμορφωθούν στην κοινωτική νομοθεσία. Αυτό νομίζω θα βοηθήσει και την Ευρώπη να πλησιάσει τον πολίτη και να έχει άμεση ε, επίδραση στις εξελίξεις στην καθημερινή ζωή και την οικονομία των κρατών μας. Το ταχύτερο, όσο το ταχύτερο γίνεται αυτό, τόσο το καλύτερο. Έληξαν εδώ οι παρεμβάσεις των βουλευτών και το λόγο θα πάρει ο Επίτροπος για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε όπως είπε η κυρία Βίγκστρομ, είναι πολύ αργά απόψε για να συζητούμε αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω πως όλοι και όλοι όσοι έλαβαν το λόγο ότι πρόκειται για σημαντικό θέμα. Ο Μάλκομ Χάρμπορ θύμισε σε τι βαθμό για τις επιχειρήσεις αυτό το ευρωπαϊκό σήμα ε, ε, ε, είναι, προσφέρει ταυτότητα εγγύηση προστατεύει και την καινοτομία και πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες μορφές προστασίας και γι' αυτό με, σε συνεργασία με την Βελγική Προεδρία θα ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα ώστε να ε, ε, ε, ολοκληρωθεί το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Σήματος ε, του Ευρωπαϊκής ε, Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να υπονομεύεται η εσωτερική αγορά. Εάν αφήναμε, αν επιτρέπαμε την υπονόμευση της ε, ενιαίας αγοράς με αυτά τα προστατευτικά μέτρα που εφαρμόνται σε κάποιες χώρες, αυτές που θα υπέφεραν τα πρώτα θύματα θα ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να πούμε stop, σταματήστε δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε παραπέρα και ευχαριστώ την κυρία μου και την ομάδα της η οποία επαγρύπνησε και έθεσε το θέμα υποβάλλοντας το σχετικό ερώτημα. Η κυρία Βίκστρομ όπως και ο κύριος Ταραμπέλα θύμισαν τι σημαίνει αυτό το κοινοτικό σήμα για τις επιχειρήσεις τη σημασία του επίσης για την ενιαία αγορά. Όπως επιθυμεί ο κύριος Ταραμπέλα, θέλω να πω ότι ακριβώς έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία αναθεώρησης για τον εξυγχρονισμό του ισχύοντος συστήματος. Η απόφαση για, για, τη, για τη δείχνει ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό, τον σχετικό κανονισμό και αυτή τη διαδικασία έχουμε ξεκινήσει με σκοπό σε αυτή την αναθεώρηση και την προσαρμογή να λάβουμε υπόψη τα σύγχρονα ε, τεχνολογικά μέσα και το διαδίκτυο και με βάση αυτό το πνεύμα θα γίνει αναθεώρηση του κανονισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Ρόιτοβα διότι ανέφερε πως είχα κάνει και εγώ τον ανταγωνισμό που θα ενταθεί εάν υπάρξει κατακαιρματισμός των σημάτων πρέπει να αντισταθούμε, πρέπει να είμαστε σε θέση να εμποδίσουμε την είσοδο προϊόντων και το πρόγραμμα δράσης θα παρουσιάσω σε λίγες εβδομάδες για την καταπολέμηση της παραποίησης θα έχει σαν σκοπό να καταρτήσει στα το... το προσωπικό ε, των κρατών μελών στα εξωτερικά σήμερα με τεχνικά μέσα για την καταπολέμηση ακριβώς της παραποίησης και της πειρατείας αλλά πρέπει να ενεργήσουμε σε διμερές επίπεδο με τα κράτη-μέλη για να μην επιτρέπουμε την είσοδο αυτών των προϊόντων. Και στο πρόγραμμα δράσης θα προβλεφθούν πιο θετικά μέτρα για τη συνεργασία με ορισμένε τρίτες χώρες, ώστε να τις βοηθήσουμε να εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική εμπορικών σημάτων και τη δική τους πολιτική καταπολέμησης της παραποίησης. Τέλος, η κυρία Χάνσλικ μου έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα. Τι θα συμβεί εάν τα εθνικά δικαστήρια επιβεβαιώσουν την απόφαση των εθνικών γραφείων καταχώρησης εμπορικών σημάτων. Βεβαίως πρέπει να περιμένουμε ποια θα είναι η αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων, να μην προδικάζουμε τίποτε. Έχω εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι θα διορθώσουν αυτά τα δικαστήρια από μόνα τους την κατάσταση. Το ενδεχόμενος μιας διαδικασίας παράβασης που αναφέρθηκε θα ληφθεί υπόψη μόνο υπό το φως των αποτελεσμάτων των προσφυγών που έχουν κατατεθεί. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε για αυτό το σημαντικό πρόβλημα που είναι και ένα από τα στοιχεία κλειδί της εσωτερικής αγοράς. Και θέλω να το πω αυτό τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε εσείς, εμείς, εσείς και σε συνεργασία με το Συμβούλιο να δώσουμε νέα ε, ε, όθηση, να τονώσουμε την εσωτερική αγορά υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολιτών. Οπότε αντιλαμβάνεστε δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε ε, οτιδήποτε που θα υπονομεύσει το ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα. Merci, Monsieur le Commissaire, le ε, έληξε η συζήτηση. 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και από τις 3 μετά το μεσημέρι έως τις 7 μετά το μεσημέρι. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες